Θα ξεκινήσουμε με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έχει ζητηθεί. Καθίστε λοιπόν. Η κυρία Φρασόνη επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, μία μικρή παρέμβαση, γιατί οι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα καθίσει όλοι. Αλλάξαμε τον κανονισμό γιατί περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο σε ανώφελες συζητήσεις και αποφασίσαμε ότι σε ό,τι αφορά την έκθεση Άουκεν ναι, δεν θα διεξαχθεί συζήτηση. Χάσαμε λοιπόν μισή ώρα μην κάνοντα τίποτα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερα αυτή την ώρα συζητώντα ένα κείμενο τόσο σημαντικό για όλου του πολίτε. Θα διαβιβάσω το σχόλιο σας στα αρμόδια όργανα. Λοιπόν, θα αρχίσει η ψηφοφορία με, την, με βάση την απλουστευμένη διαδικασία έκθεση Κλάους Λένε σχετικά με τη Λευκή Βίβλο, σχετικά με τις αγωγέ αποζημίωση για παραβίωση της αντιμονοπολιακής νομοθεσίας. Αρχίζει η ψηφοφορία, μία ψηφοφορία θα γίνει. Ψηφίσατε όλοι. Πραγματικά ψηφίσατε όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. Λοιπόν, 526, 498 υπέρ, 11 κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Λέν. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη, έχουμε έκθεση Σικέρσκη, διανομή τροφίμων στους απόρους. Θεωρώ ότι νομίζω ότι ο εισηγητής θέλει στα γρήγορα να πάρει το λόγο. Szanowni posłowie, przyjmując dzisiejszy raport dotyczący programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej αφορά την διανομή τροφίμων στους άπορους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να δώσουμε το σωστό μήνυμα προς τους πολίτες μας <clears throat> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει αυτούς οι οποίοι είναι ενδεείς και χρειάζονται αρρωγή με την δωρεάν διανομή τροφίμων. Προγράμματα όπως αυτό το είδος, όπως η διανομή φρούτων στα σχολεία αλλάζουν και τη συνολική αντίληψη που έχουν οι πολίτες μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει πιο φιλική την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη αρρωγής και ιδίως τους νέους. Η έγκριση αυτής της έκθεσης θα καταδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοντά στους πολίτες. Ευχαριστώ τώρα. Θα σε συζητήσω με την πρόταση ψηφίσματος τροπολογίες της Αρμόδιας Επιτροπής συνολικά. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άρθρο 27, παράγραφος 2, 2, 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση ηλεκτρονική. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2,29 υπέρ, 308 κατά. Περνάμε στο 14 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 27 παράγραφος 7, 16 έως 29 τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, μερικοί δεν κούνησαν καν το χέρι τους. Έναρξη ψηφοφορίας, επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας σαφώς εγκρίθηκε. 361 υπέρ, 177 κατά, 6 εποχές. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται να σε επαληθεύσουμε. Επαλήθευση για την τροπολογία 5. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας. 379 υπέρ, 171 κατά. Λοιπόν, πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές. Ε, συγχαρητήρια κύριε Σικάς. Α, παραμένει το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε σαφώς, 425 υπέρ, 71 κατά, 62 αποχές και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Οπότε, έκθεση ε, Καρίμα για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Ε, έχουμε ε, την ονομαστική ψηφοφορία για την πρώτη ονομαστικού ψηφίσματος 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 326 υπέρ, μείον 226, δηλαδή 100 λιγότεροι, τρεις αποχές. Το υπόλοιπο καταπίπτει, τροπολογία υπαριθμών 1 με ονομαστική. Α, καταπίπτει. Περνάμε στο επόμενο θέμα, γιατί όλα αντικαθίστανται από αυτά που εγκρίναμε. Έκθεση Λέτινεν για την κοινωνική ε, ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων σε αλυσίδε παραγωγή. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματο. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να απολυθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 231 υπέρ, 303 κατά. Περνάμε στο 2, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 321 υπέρ, 235 κατά, 11 αποχές, εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα λοιπόν καταπίπτουν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σύμφωνα με την ομερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση Κατερίνας Μπατζελή για τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, το λόγο έχει η εισηγήτρια, κυρία Μπατζελή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κύριε Πρόεδρε να υπήρχε δυνατότητα σύγκρισης του ψηφίσματος της έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και του εναλλακτικού ψηφίσματος των 40 μελών και του Άλντε. Θα διαπίστωνε πρώτον ότι τροποποιούνται συνολικά 15 προτάσεις χωρίς να δίνουν ένα μήνυμα δεύτερο πέρα του ποσοτικού υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα όπου η εναλλακτική πρόταση διαγράφει κάθε αναφορά του ρόλου και της ευθύνης των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων λιανικής και χονδρικής πώλησης. τρίτον αυτοακυρώνεται η γραπτή δήλωση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με τις 439 υπογραφές συναδέλφων όπου θέλουν τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία των σούπερ μάρκετ και τέταρτον διαγράφεται ή εξοραίζεται κάθε πολιτική αθέμητου ανταγωνισμού ενώ ακόμα φτάνει ακόμα και στην άρνηση της σύστασης δημιουργίας πανευρωπαϊκής δράσης δεδομένων για τις τιμές παραγωγού καταναλωτή προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες και καταναλωτές. σκοπός της επιτροπής γεωργίας αλλά και της ομάδας υψηλού επιπέδου είναι να εξεταστούν οι πρακτικές του ανταγωνισμού και η διαφάνεια της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τροφίμων. σήμερα όλοι κρινόμαστε. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου με δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Η κυρία Λούλινγκ, διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους ότι είμαι ένα από τους συντάκτες της του εναλλακτικού ψηφίσματος. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στη Σοβιετική Ένωση. Είμαι σίγουρος αγαπητοί συνάδελφοι ότι όλοι γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί έδωσα το λόγο στην ε, ε, εισηγήτρια, έχει δικαίωμα να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Έγινε σεβαστή απλώς η ελευθερία του εισηγητή. Δύο τροπολογίες. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 131 ΕΠΕΡ, 399 κατά, 39 αποχές απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα της Αρμόδιας Επιτροπής, ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 573, 390 υπέρ, 112 κατά, 71 αποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Πατσελή. Η μερσία διάταξη προβλέπει τη ψηφοφορία της έκθεσης Άουκεν για τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία. Ο κύριος Κάσμαν που θα ήθελε να κάνει μια σύντομη δήλωση. Ο κύριος Κάσμαν. Όχι, ο κύριος Κάσμαν πρώτα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Όκεν, ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι για λόγους αρχής θα ήθελα να αποσυρθεί το όνομά μου από το ενακτικό ε, ψήφισμα της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Θα επιθυμούσα να σας γνωστοποιήσω ότι μετά από πέντε χρόνια ανασχόλησης με αυτό το θέμα θα ψηφίσω κατά και των δύο εναλλακτικών προτάσεων ψηφίσματος και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Άουκεν. Ευχαριστώ. Merci pour cette précision. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ο εισηγητής. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα της ε, εργασίας των μελών της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Ως εισηγήτρια πάντοτε κατέβαλα προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα που επηρέασε πάρα πολύ την ε, ζωή πολλών πολιτών που ζουν στην Ισπανία. Επηρέασε επίσης και το περιβάλλον και την οικονομία στην Ισπανία. Η έκθεση είναι η έκθεση της Επιτροπής, υιοθετήθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο ε, κάνει διάκριση μεταξύ διαφόρων πτυχών του φαινομένου της ε, αστιφιλίας στην Ισπανία. Εδώ αναφέρεται το θέμα των βασικών δικαιωμάτων των Ευρωπών πολιτών στην ιδιοκτησία και όλες οι χώρες μέλη δεσμεύονται από αυτό. Το πρόβλημα των αρνητικών επιπτώσεων της ε, φιλία, στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές και στα Ισπανικά νησιά αλλά και αλλού είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από την ε, Μαδρίτη. Υπάρχει το πρόβλημα της επαναφοράς του νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε το 1988 πράγμα που θα συμβαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς σπίτι αφού τα σπίτια τους θα καταδαφιστούν. Το θέμα της επίπτωσης που έχουν οι παράνομες κατοικίες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ συχνά υπάρχουν αθώοι αγοραστές που είναι θύματα όλων αυτών των διαδικασιών της αστιφίλειας. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το που βρίσκεται η ευθύνη για όλες, για όλα αυτά τα προβλήματα και θα λυπάμαι για τις παράνομες δράσεις των αρχών γιατί πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο πλήττει την αηφόρο ανάπτυξη καθώς και την προσπάθεια για διασφάλιση, ε, για προστασία του περιβάλλοντος. Στην έκθεση αυτή θα έπρεπε να τύχει μια πλήρου ε, συζήτηση. Οι κανόνε αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ιδιαίτερα όταν οι εκθέσει που αφορούν αναφορέ από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχουν άμεση σχέση με αυτό. Θα ήθελα να απορρίψω και τι δύο εναλλακτικά ψηφίσματα. Πιστεύουμε ότι δεν αντικατοπρίζουν τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από πλευράς Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πολύ. Επί του συνόλου του κειμένου υπάρχουν δύο τροπολογίες. Έχει αποσυρθεί το αίτημα για νομαστική ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία, να κάνουμε επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Όπως Φαντάστηκα, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Όχι. Δεν θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. και χθε σύμφωνα με τον κανονισμό. Τροπολογία 2, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Επαλήθευση. Ωραία. Ωραία να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Πιστεύω ότι το είχα καταλάβει καλά. 436 κατά, 72 υπέρ, 44 αποχές. Συνεπώς απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα της Αρμόδιας Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψήφισαν 573, 349 υπέρ, 110 κατά, 114 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Άουκεν. Ακολουθεί η έκθεση Μίλαν Μόνς για τις διατλαντικές σχέσεις μετά από τις προεδρικές εκλογές στο Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Τροπολογία 4. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 240 υπέρ, 307 κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 19. Χωριστή ψηφοφορία, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 με, σε τμήματα, σε τρία τμήματα με ονομαστική κλίση για όλα τα τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 97 υπέρ 465 κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 483 υπέρ, 48 κατά. 37 αποχές τελευταίο τμήμα, άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 259 υπέρ, 290 κατά, με μικρή πλειοψηφία, απορρίπτεται και το τρίτο τμήμα. Τροπολογία 36 με χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 41, τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται θα το ελέγξουμε. Δεύτερο βήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Τι να τους κάνω. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Με μεγάλη πλειοψηφία απερίφθη. Παράγραφος 45 με χωριστή ψηφοφορία. Υπέρο. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 52, τροπολογία 6, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοθυρίας. 72 υπέρ, 472 κατά 11 αποχέ. Το σύνολο του ψηφίσματο όπω τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 503 υπέρ 51 κατά 10 αποχές με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Μίλαν Μον. Δύο προτάσεις ψηφίσματος για την, εμπορική, την ενδιάμεση εμπορική σχέση, συμφωνία με το Τουρκμενιστάν. Δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Κάσπαρη για, ένα διαδικαστική, για διαδικαστική παρέμβαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βάσει του άρθρου 174 η ομάς του ΕΛΚ ζητά η τελική ψηφοφορία να αναβληθεί για την επόμενη Ολομέλεια. Στη χθεσινή συζήτηση ήταν φανερό ότι μια πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει παρά τις αμφιβολίες της αυτήν την συμφωνία. πολύ συνάδελφοι θεωρούν ότι με αυτή τη συμφωνία μετά από πολλά χρόνια δράνης θα περάσουμε σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο στη σχέση με το Τουρκμενιστάν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην λάβουν λαθασμένα μηνύματα το Συμβούλιο και η Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρξει αμφιβολία ότι σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να θεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία. Δυστυχώ, η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν δεχτήκανε καθόλου αυτήν την αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσω του συναδέλφου μου να αναβάλουν την τελική ψηφοφορία μέχρι ότου το Συμβούλιο και η Κομισιόν δεχτούν το αίτημα του Κοινοβουλίου. Βάσει του άρθρου 174 του κανονισμού μας λοιπόν, έχει εκφραστεί λοιπόν η άποψη μιας πολιτική ομάδος. Ζητώ αν υπάρχει ένα ομιλητή υπέρ και ένα ομιλητή κατά αυτή τη πρόταση. Υπέρ, ο κύριο Βίσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μας τον κύριο Κασπάρη ότι πρέπει να αναβάλουμε την τελική ψηφοφορία <clears throat> για την έκθεση αυτή γιατί ήταν σαφές από τη χθεσινή συζήτηση ότι ιδίω στο Συμβούλιο και σε μικρότερο βαθμό η Κομισιόν δεν ήταν έτοιμοι να δώσουν στο Ευρωπαϊκό, το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να έχει μια ενδελεχή παρακολούθηση της κατάστασης στο Τουρκμενιστάν και εφόσον δεν έχουμε επαρκείς εγγύησης από το Συμβούλιο, υποστηρίζουμε και εμείς στο Σοσιαλιστικό Κόμμα τη θέση του κ. Κασπάρη και την αναβολή της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εκφραστεί κατά? Εάν όχι, θέτω σε ψηφοφορία την αίτηση ε, αναβολής ψήφι υπέρ, κατά, απόχες. Αναβάλλεται λοιπόν η τελική ψηφοφορία για τα θέματα αυτά. και η έκθεση Κασπάρη για τον ίδιο λόγο αναβάλλεται η... Κύριε Κασπάρη, ναι, έχετε το λόγο και πάλι. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, μόνο για την τελική ψηφοφορία ζητήσαμε να γίνει η αναβολή, όχι για την ψηφοφορία σε σχέση με τις τροπολογίες. Α, δεν είχα πάρει σωστές πληροφορίες. Μόνο η τελική ψηφοφορία θα αναβληθεί. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες όμως. Έχουμε επομένω την έκθεση Κάσπαρη σε σχέση με την ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν. Έχουμε τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και σταματάμε εκεί. Έχουμε τώρα την έκθεση Λαμπρινίδη για την ενίσχυση των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο. Σα παρακαλώ κύριε Κασπάρη. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρο. Σας ζήτησα να αναβάλλετε τις δύο τελικές ψηφοφορίες αλλά να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες. Μόνο τις τελικές ψηφοφορίες να αναβάλουμε, όλες τις άλλες τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε. <clears throat> Εντάξει. Η γραμματεία μας δεν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για αυτό. Εγώ είχα καταλάβει θα ψηφίζαμε τις τροπολογίες για το Τουρκμενιστάν, όχι για τη δική σας. Ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων, ε, τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Παράφος 2, τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά, απόχες, απορρίπτεται. Η παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές Τι Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. 297 υπέρ, 256 κατά, 6 αποχές, γίνεται δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγωση 5, τροπολογία 1, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 2.38 υπέρ, 311 κατά, 8 αποχές, απορρίπτεται. Ακολουθεί τροπολογία 5 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Με προφορική τροποποίηση κυρία Φλότρο. Η τροπολογία αυτή της ομάδας μου επιτρέπει να ασχίσουμε πίεση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βελτιωθεί αν αντικαταστήσουμε την έννοια της προοπτικής υπογραφής μιας συμφωνίας με την προοπτική της περάτωσης της διαδικασίας κύρωσης αυτής της συμφωνίας που είναι η σωστή διατύπωση. Μάλιστα. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι κατά αυτής της τροπολογίας προφορικής. Δεν βλέπω 40 συναδέλφους να έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους. Θέτουμε λοιπόν σε ψηφοφορία αυτή την παράγραφο όσο έχει τροποποιηθεί προφορικά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφεται. Θα ελέγξουμε τροπολογία 2, έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε σα τα είχα πει. 147 υπέρ, 386 κατά, 16 αποχές είχε απορριφθεί. Τροπολογία 7 στην παράγραφο 8. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και δεν θα φτάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία διότι έχει αναβληθεί για την επόμενη ολομέλεια. Κατάλαβα αυτά που θέλει να πει ο εισηγητής μας λοιπόν. Σύμφωνα με την μίληση διάταξη θα ψηφίσουμε για την έκθεση του κύριου Λαμπρινίδη για την ενίσχυση της ασφάλειας. Α, κύριε Γκέμπελ, έχετε το λόγο. Πρόβλημα πάλι. Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι ζητήσατε ψηφοφορία για την έκθεση Κάσπαρη και ότι η τροπολογία της ε, Ομάδα μου καταψηφίστηκε. Εγώ ίδιο το καταψήφισα γιατί ανακατεύτηκε η σειρά. Σα ζητώ να επαναληφθεί. Μία τροπολογία είχατε πει και μετά δεν θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Καταρχήν, στις οθόνες φαινόταν αυτό το οποίο έλεγα. Αν όμως οι συνάδελφοι επιθυμούν να ξαναγίνει ψηφοφορία γι' αυτό, πολύ ευχαρίστως. Δεν θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, ένα λεπτό να επιστρέψω στο φάκελο. Τροπολογία 1 της σοσιαλιστικής ομάδας λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται πράγματι. Αυτό αλλάζει την κατάσταση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη επιτέλους Φτάσαμε στην ψηφοφορία που ανακοίνωσα τρει φορέ, έκθεση Λαμπρινίδη, ενίσχυση ασφάλεια και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο. Ε, τώρα, ε, θα εξετάσουμε την έκθεση προτάσεων. Παράγραφος 1, μετά το H. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική. Έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 2.21 υπέρ, 3.17 κατά, 9 αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται σε επαλήθευση. Επαλήθευση για την τροπολογία υπαρθμών 4. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.29 υπέρ, 2.79 κατά, 24 αποχές. Τροπολογία 5, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 2.44 υπέρ, 2.91 κατά, 5 αποχές απορρίπτεται. Νομίζω ότι το ΕΛΚ θέλει να υποβάλει ε, προφορική τροπολογία. Σωστά νομίζω. Υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ. Α, δεν με ενημέρωσαν σωστά από ό,τι φαίνεται. Σας επισημαίνω ότι για πρώτη φορά βρίσκονται οι γονεί μου στο, ε, στην ε, αίθουσα και σήμερα μου δημιουργείται δυσκολίες. Τέλος του διαδικαστικού. Παράγραφος 1, τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε παράγραφος 1. Χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολλοί συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Επαλήθευση αναγκαστικά. Παράγραφος 1. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Πολύ σωστά. Κάναμε και επαληθεύσαμε 2,51 υπέρ, 260 κατά, 8 αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, αιτιολογική σκέψη Q Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σύνολο της πρώτης ονομαστικού ψηφίσματος αποστροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία έναρξη. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 4,81 υπέρ, 25 κατά, 21 αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τελευταία λοιπόν ψηφοφορία. Α, ο εισηγητής, ο κ. Λαμπρινίδης, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευγνώμων για όσους υποστήριξαν. Μία σύγχυση. Η η προφορική τροπολογία υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφοριών, αλλά κανένα δεν υποστήριξε. Υποθέτω ότι καταπίπτει, έτσι δεν είναι, αφού δεν ψηφίστηκε. Σωστά, εντάξει. Πράγματι, σα επιβεβαιώνω ότι για να εγκριθεί μία προφορική τροπολογία πρέπει προφορικά να εκφραστεί, δεν συνέβη αυτό. Τέλος, πρόταση ψηφίσματος ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων. Παράγραφος 3, τροπολογία 1, υπέρ κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται αλλά επαλήθευση. Ε, νομίζω απορρίπτεται αλλά επαλήθευση, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται 229 υπέρ, 264 κατά, 4 αποχές. Παράγραφος 3 χωριστή ψηφοφορία υπέρ. Κατά εγκρίνεται αυτή. Παράγραφος 14 χωριστά. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι το δεύτερο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2,82 υπέρ, 2,15 κατά. Το 15 με χωριστή ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη, ψηφίσατε, πέρας ψηφοφορίας. 4,69 υπέρ, 8 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται, συγχαρητήρια στους συντάκτες. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες, αλλά αρχίζουν ε, οι επεξηγήσεις ψήφου.